Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση, η διακοπήσα. Τα πρακτικά τη χθεσινή όσο είναι στη διάθεσή σα. Έχετε παρατηρήσει όσον αφορά τη χθεσινή συνεδρίαση και τα πρακτικά τη. Όχι, εν τη αυτή περιπτώσει θεωρούνται συγκεκριμένα τα πρακτικά. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο.